Τελευταία ανακοίνωση. Βάσει του άρθρου 211 παράγραφος 3 η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων προτείνει την εξής ερμηνεία του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις υποψηφιότητες και τις ε, γενικές διατάξεις. Εάν πρέπει να αντικατασταθεί μόνο ένας αντιπρόεδρος ε, και υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, μπορεί να, ελεχθεί, ε, να εκλεγεί διαβοής. Ο πρόεδρος έχει τη διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσει αν θα γίνει ψηφοφορία μέσω ε, μυστικής ψηφοφορίας ή διαβοής ο υποψήφιος ε, που εκλέγεται ε, παίρνει τη θέση του αντιπροέδρου που αντικαθιστά. Εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση στη συγκεκριμένη ερμηνεία μέχρι αύριο, τη 23 Ιουνίου, θα θεωρήσουμε ότι αυτή η ερμηνεία εγκρίνεται.